Colleagues, colleagues, let Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα πρέπει να σεβαστούμε τις χρονικές προθεσμίες τις οποίες έχουμε. Ο Επίτροπος θα πρέπει να φύγει στις 12.30 ακριβώς. Συνεπώς έχουμε 65 λεπτά στην διάθεσή μας και γι' αυτό παρακαλώ θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι στις ερωτήσεις τις οποίες θα θέσετε, εξαιρετικά σύντομοι. Θα συζητήσουμε επί μακρόν τις εκθέσεις αναχώρα όταν είναι έτοιμες. Σας θυμίζω ότι θα τα συζητήσουμε αυτά. Και γι' αυτό παρακαλώ να σεβαστείτε ε, τον χρόνο και να είσαστε πάρα πολύ συνοπτικοί και θα, θα είμαστε πολύ αυστηροί. Βλέπω όσους ζήτησαν το λόγο, τους βλέπω λέει ο Πρόεδρος. Τους, τους βλέπω λέει ο Πρόεδρος αυτούς που έχουν ζητήσει το λόγο. Έτσι κι αλλιώς ε, οι συγητές από τη μία και οι α, ε, συντονιστές από την άλλη ε, θα πάρουν αυτόματα το λόγο αν θέλετε. Ο κόσμος αλλάζει, συνάδελφοι. Έχετε για διαδικαστικούς λόγους τον λόγο. Κύριε Μποργέζιο, για διαδικαστικούς λόγους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εδώ, να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίηση της πολιτικής μου ομάδας για το αποτέλεσμα στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, όπου εξελέγει ένας μεγάλος πατριώτης. Ζήτω οι πατριώτες όλου του κόσμου. Κοιτάξτε, σέβομαι τις προσωπικές σας απόψεις, αλλά παρακαλώ κρατήστε για τον εαυτό σας. Δεν είναι η στιγμή και η ώρα να το συζητήσουμε, είστε εκτός θέματος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, λέει ο κύριος Πάσκου, ο κόσμος αλλάζει, αλλάζει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Θα πρέπει να παραμείνουμε στον δρόμο που έχουμε επιλέξει. Και γι' αυτό αμέσως θα ζητήσω από τον Επίτροπο Χάν να μας κάνει την εισαγωγική του παρέμβαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει τόσο πολύ που ξεκινάμε ίσως και νωρίτερα από τον χρόνο τον οποίο προεβλέπετο, λέει ο Επίτροπος. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει στον τομέα της διεύρυνσης. Πέρυσι είχαμε πει ότι θα καλύψουμε σε επίπεδο μεσοπρόθεσμης στρατηγικής θα κάνουμε μια επισκόπηση της προσπάθειας την οποία κάναμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Γιούνκερ ενώ και θα πούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι χώρες ε, οι οποίες έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Οι χώρες συνεχίζουν την προσπάθεια, συνεχίζεται η προσπάθεια επίσης και για τον εξυγχρονισμό της νοτιοανατολικής Ευρώπης και αυτό δημιουργεί ασφάλεια θα έλεγα ένα αξιόπιστο περιβάλλον για τις χώρες μας και τις γειτονικές χώρες και ε, η διεύρυνση σε κάποια φάση είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πράγματα προχωρούν, προχωρούν με ανησυχητική ταχύτητα σε ορισμένες περιπτώσεις όμως και κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν περίπλοκα προβλήματα και διαρθρωτικές δυσκολίες. Η κατάσταση λοιπόν είναι δύσκολη, θα πρέπει εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολλές είναι οι χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει σοβαρές προσπάθειες να ανακαινήσουν σε εισαγωγικά τα νομικά του συστήματα και τα δικατικά συστήματα. Η Αλβανία υιοθέτησε συνταγματικές τροπολογίες τον Ιούλιο που θα είναι η βάση για την δικαστική μεταρρύθμιση. Πολλές χώρες όμως, πολλές είναι οι χώρες όπου το δικαστικό σύστημα δεν έχει την απαιτούμενη ε, ανεξαρτησία και αυτονομία. Τα τελευταία χρόνια οι χώρες έχουν καθορίσει τα πλαίσια τους, ανακαθορίσει τα πλαίσια τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι πολιτικές αυτές αποφάσεις θα πρέπει να γίνουν πραγματικά αποτελέσματα. Ε, θα πρέπει να καθοριστούν οι συνθήκες ε, κάτω από τις οποίες θα γίνουν ε, οι προσπάθειες αυτής, θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα εγκληματικά δίκτυα, η τρομοκρατία που συνιστά απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ίδιες τις χώρες διεύρυνσης. Απαιτείται περαιτέρω συνεργασία τα θεμελιώδη δικαιώματα θα συνεχίσουν να εδράζονται στο κράτος δικαίου, αλλά σε επίπεδο όμως πρακτικής εφαρμογής εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες και σε επίπεδο μέσων ε, ενημέρωσης, σε επίπεδο ελευθερίας έκφρασης, σε επίπεδο ε, διακρίσεων εις βάρος συγκεκριμένων ε, εθνοτικών ομάδων Υπάρχουν διαφοράς, διαφορές βέβαια ανάμεσα στις χώρες. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί εδώ ο κεντρικός ρόλος που παίζει το, ο κοινοβουλευτικός βραχίωνας της ε, προσπάθειας αυτής και κάποιες ε, πολιτικές αντιλήψεις οι οποίες διαιρούν και δεν ενώνουν θα πρέπει να ξεπεραστούν. Έχουμε εμείς ανανεώσει τους τρόπους στήριξης προς τις χώρες αυτές έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι χώρες διεύρυνσης αντιμετωπίζουν όμως προκλήσεις κοινωνικές, διαφθρωτικές, οικονομικές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους το κράτος δικαίου και οι τρόποι σεβασμού του κράτους δικαίου δημιουργούν μερικές φορές ε, καταστάσεις δύσκολες. Εγώ σας παρουσίασα μια εικόνα εσκεμένα, θα έλεγα, ε, αντικειμενική σε εισαγωγικά. Ε, κανένας δεν μπορεί να υπογραμμίσει το μέγεθος της διαδικασίας αυτής στρατηγικής διεύρυνσης και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούν δεδομένο οι ηγεσίε των χωρών μας. Θα πρέπει να πούμε και στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η πολιτική αυτή είναι ζωτική για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στα πλαίσια της μεταναστευτικής κρίσης αυτό αποδεικνύει θα έλεγα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μην είναι παρούσα στον τομέα της γεωπολιτικής της παρουσίας. και ξέρουμε τα βήματα τα που έχουν γίνει στον τομέα του λεγόμενου διαδρόμου της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, τη συμφωνία με την Τουρκία. Ξέρουμε τα αποτελέσματα μείωση των θανάτων στην θάλασσα, στην περιοχή αυτή, όπως επίσης και μείωση του αριθμού των ανθρώπων που μεταναστεύουν ή που πηγαίνουν σαν πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά κάποια φάση είχαμε φτάσει ε, ε, ε, τα 740.000 μετανάστες και πρόσφυγες που είχαν περάσει μέσα από τα ελληνικά νησιά και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που ακολούθησε ο αριθμός αυτός έπεσε σε πραγματικά πολύ χαμηλά επίπεδα. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι είναι, υπάρχει ακόμα θέμα, ότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί, αλλά παρόλα αυτά αυτοί που πιστεύουν ότι η κρίση αυτή έχει τελειώσει και που θεωρούν ότι μπορούμε να πούμε business as usual, αυτό δεν ισχύει. Και θα πρέπει να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύει όλες τις χώρες στην καταπολέμηση των συστημάτων αυτών δουλείας τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Δεν θα πρέπει φυσικά να κρατήσουμε στα σύνορα τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης προχωρούμε και σε άλλους τομείς όπως την λεγόμενη ατζέντα στον τομέα της συνδεξιμότητας. Αυτό το connectivity agenda συνδέει τους ανθρώπους, τις χώρες, τις υποδομές Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή και έτσι θα δημιουργήσουμε όχι μόνο οικονομικές δυνατότητες αλλά θα βελτιώσουμε και τις αγαστές γειτονικές σχέσεις. Τέλος, αγαπητά μέλη, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια σημεία αναχώρα. Θα ξεκινήσω με την Τουρκία. Εμείς είμαστε κομβικοί εταίροι μεν τον δε με την χώρα αυτή αυτό το οποίο έγινε τον Ιούλιο το πραξικόπημα ήταν ε, μια επίθεση στη δημοκρατία. Ήμασταν οι πρώτοι που το καταδικάσαμε και έπρεπε να υπάρξει ανταπάντηση. Ήταν θεμητή η ανταπάντηση. Αλλά η μεγάλη εμβέλεια των μέτρων τα οποία λαμβάνονται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες μας ανησυχεί. Η Τουρκία σαν υποψήφια χώρα θα πρέπει να πληρεί τα υψηλότερα επίπεδα σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχει αναλάβει την υποχρέωση να το κάνει και πάνω σε αυτό δεν μπορεί να υπάρχουν παραχωρήσεις. Συνεπώς στην φετινή έκθεση εμείς σημειώνουμε την υπαναχώρηση του σεβασμού της Τουρκίας στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα μέτρα τα οποία ελήφθηκαν από τον Ιούλιο μέχρι και αυτά που ελήφθηκαν τις τελευταίες, ελήφθησαν τις τελευταίες μέρες δείχνουν ότι δεν είναι σαφής ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν μέτρα καταστολής τα οποία λαμβάνονται και απέναντι στους Κούρδους και όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ελευθερίας έκφρασης. Τα μέτρα φύγουν το σύνολο της κοινωνίας, την αστυνομία, τις αρχές καταστολής, το στρατό, τα μέσα ενημέρωσης, η φυλάκιση των, της ηγεσία του ΧΑΝΤΕΠΕ την προηγούμενη εβδομάδα είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και δείχνει ότι η κατάσταση στο νότιο ιδιαίτερα τμήμα της χώρας είναι πολύ ανησυχητική. Και επίσης κάποιες απειλές για την επαναφορά της θανατικής ποινής είναι πράγματα ασύμβατα με την επισήμως εκφρασμένη επιθυμία της Τουρκίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά εμείς δείχνουμε μια κάποια κατανόηση απέναντι σε μια ισχυρή απάντηση στην απειλή του πραξικοπήματος και αναγνωρίζουμε και τα βήματα προόδου και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο ε, οικονομικό τα τελευταία χρόνια. Πρέπει όμως η Άγκυρα να αποφασίσει τι θέλει. Έχει να περάσει ένα τεστ αξιοπιστίας απέναντι στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά έχουμε εμβαθύνει σε τέσσερις τομείς κοινού συμφέροντος την συνεργασία και μετά από την συνάντηση της 29ης Νοεμβρίου του 2015, συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καταρχάς, δώσαμε μια ισχυρή οικονομική βοήθεια για την, για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Η Τουρκία στον τομέα επίσης έχει και ανέβει σε επίπεδο σε σχέση με ε, την χορήγηση θεωρήσεων. Είχαμε αναλάβει εμείς την υποχρέωση ε, να απελευθερώσουμε το καθεστώς των θεωρήσεων εφόσον η Τουρκία είχε εκπληρώσει το σύνολο της διαδικασίας. Προχωρήσαμε στο άνοιγμα επίσης δύο επιπλέον κεφαλαίων ε, στο τέλος του 2015 και στις αρχές του 2016. Ε, νομίζω ότι οι σχέσεις μας ε, ε, μπορούν να είναι σε ένα επίπεδο πολύ δραστήριο και σοβαρό. Αυτά για την Τουρκία. Τώρα για το Μαυροβούνιο ή τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο με τις εκλογές του Οκτωβρίου οι οποίες έγιναν με πιο διαφανή και συμμετοχικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν υπήρξε πλήρης σεβασμός από ό,τι φαίνεται του κράτους δικαίου. Το σύστημα όμως τώρα θα πρέπει να δουλέψει, <clears throat> θα πρέπει να υπάρξει η δικαστική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα <clears throat> στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η Σερβία επίσης ε, πήρε μέτρα, άνοιξαν τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια και στα πλαίσια της εσωτερικής πολιτικής και στα πλαίσια των σχέσεων με το Πέδιο. Η πορεία των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί από την πρόοδο σε όλους αυτούς τους τομείς και η Σερβία έχει φυγεί από την μεταναστευτική κρίση και έπαιξε ένα επικοδομητικό γενικά ρόλο. Οι οικονομικές προσπάθειες έχουν ε, δώσει αρκετά αποτελέσματα για τη ΦΥΡΟΜ δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από την εσωτερική πολιτική κρίση παρά το ότι τον τελευταίο καιρό έγιναν κάποια βήματα. Υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να ξεπεραστεί η συστημική κρίση. Πρέπει να υπάρξει ε, μια σωστή διαδικασία για τη διοργάνωση των εκλογών όπως η Σερβία έπαιξε ρόλο σημαντικό για την καταπολέμηση της μεταναστευτικής κρίσης και συνεργάστηκε με τις γειτονικές χώρες και τα κράτη-μέλη. Υπό το φως αυτής της πορείας λοιπόν εμείς εξακολουθούμε να εμένουμε στις συστάσεις μας για την κίνηση των διαπραγματεύσεων αλλά <clears throat> οι προϋποθέσεις που υπήρχαν και πέρυσι σε σχέση με ε, την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών παραμένουν. Η Αλβανία συνεχίζει και αυτή να κάνει σταθερή πρόοδο για την εκπλήρωση των πέντε αρχικών προτεραιοτήτων έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι οι συνταγματικές τροπολογίες οι οποίες έγιναν ομόφωνα δεκτές <clears throat> τον Ιούνιο του 2015 θα επιτρέψουν να υπάρξει μια πλήρης αναθεώρηση και της λειτουργίας του δικατικού συστήματος και της δημόσιας μηχανής. οι διαδικασίες ε, καταπολέμησης ε, ε, απέναντι στην διαφθορά, της διαφθοράς μάλλον, του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει να συνεχιστούν και να εμβαθυνθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εδώ Δίνουμε λοιπόν μια σύσταση υποαίρεση εφόσον συνεχιστούν οι προσπάθειες ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης ιδιαίτερα σε σχέση και με την λήψη υπόψη του ρόλου των υπολείπων κοινωνικών παραγόντων της χώρας όπως εκκλησίες κτλ. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει κάνει και αυτή σημαντικά βήματα προόδου. Αυτό επιτρέπει σε μας να γνωμοδοτήσουμε απέναντι στο αίτημα Οι ηγέτες της χώρας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα βαθύτατα διαφορετικά προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας, να ενισχύσουν το κράτος δικαίου, να ενισχύσουν τη δημόσια διοίκηση, την βελτίωση της ε, κυβερνησιμότητας της χώρας. Όλες αυτές είναι προτεραιότητες που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Για το κοσυφοπέδιο η Συμφωνία Σταθεροποίησης η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία πλέον παρέχει το απαιτούμενο πλαίσιο για στενές οικονομικές σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα αυτή έχει κάνει σημαντικά βήματα για την εκπλήρωση των προποθέσεων του οδικού χάρτη για τη χορήγηση των θεωρήσεων και στα πλαίσια των προτάσεων που έγιναν τον Μάιο του 2016 έχουν υπάρξει θετικές συστάσεις για το σύστημα θεωρήσεων. Ε, η, η πολιτική αυτή στασιμότητα όμως ε, η οποία σημειώνεται στην Πρίστινα θα πρέπει να ξεπεραστεί γιατί έχει συνέπειες στις διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και στον σεβασμό του κράτους δικαίου. Αγαπητοί ε, φίλοι, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της έκθεσης για φέτος. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν είναι αυτός Είναι ένα στρατηγικό μέσο έτσι ώστε να προχωρήσουν οι οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι κάτι που θέλει χρόνο, είναι κάτι που είναι δύσκολο, αλλά κάθε βήμα που γίνεται, κάθε benchmark που επιτυγχάνεται είναι κάτι που βελτιώνει την ανθεκτικότητα και την ενίσχυση της σταθερότητας στην άμεση γειτονία μας. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν την πολιτική αυτή. Εγώ βέβαια δεν θέλω να επιβάλλω λύσεις. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες των προτάσεων αυτών. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι η αίσθηση στις χώρες αυτές ότι οι διαδικασίες αυτές είναι κυρίως δικές τους και είναι υπεύθυνοι για αυτές. Θα πρέπει να κάνουν λοιπόν τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτείται έτσι ώστε τα συστήματα και τα μέσα που θα οδηγήσουν στην διεύρυνση να θεωρηθούν ότι τους ανήκουν. Πολλές από τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν στις χώρες διεύρυνσης. Κοιτάξτε, τα Δυτικά Βαλκάνια βλέπετε στον χάρτη είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεωγραφικά. Είναι συμφέρον του καθενός μας και όλων μας να σταθεροποιήσουμε την περιοχή ακόμα περισσότερο. Υπολογίζω λοιπόν στην ισχυρή και συνεχιζόμενη συνδρομή σας στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τις χώρες διεύρυνσης. Η συνεισφορά σας είναι κομβική, ιδιαίτερα σε σχέση με τον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω για δύο χρόνια στενής και εξαιρετικής συνεργασίας. Πολλοί από εσά μεμονωμένα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο ασχολούμενοι με μία χώρα ξεχωριστά ο καθένας και νομίζω ότι η επιτυχής πρόοδος που έχει γίνει οφείλεται και σε εσά. Εδώ θα απευθύνομαι και στους συναδέλφους από τα μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους συμπολίτε μας στις διάφορες χώρες για την ανάγκη αυτής της συνέχισης αυτής της διαδικασίας και να μιλήσουμε για τις θετικές συνέπειες των μέτρων τα οποία λαμβάνονται προς όφελος της Ευρώπης, του συνόλου της Ευρώπης, ιδιαίτερα στον τομέα της σταθεροποίησης των άμεσων περιοχών γειτονίας μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Έχουμε 44 λεπτά και μετά θα πρέπει να φύγει ο Επίτροπος και έχουμε πολλούς ε, συναδέλφους ε, που θέλουν να παρέμβουν για να σχολιάσουν ή να υποβάλουν ερωτήσεις. Ε, δεν χρειάζεται να διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κανόνας τον οποίο θέλετε να, το οποίο θέλω να εγκρίνετε έχει ως εξής. Αυτοί που είναι εισηγητέ και συντονιστές θα μιλήσουν για δύο λεπτά. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι είτε εισηγητέ είτε συντονιστές, αλλά όχι και τα δύο, θα μιλήσουν για ένα λεπτό. Παρακαλώ να τηρήσετε αυτό τον κανόνα, γιατί προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να προλάβουμε. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Ο κύριος είναι ο κύριος Πρέντα. Καταρχήν κύριε Επίτροπε θα ήθελα να σας συγχαρώ για την έγκριση του πακέτου του διεύρυνση του 2016. Θεωρώ ότι είναι πράγματι σημαντικό να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές σας όσον αφορά την εξέλιξη της μεθοδολογίας της διεύρυνση, αλλά και επίσης να ε, υλοποιηθούν οι παρουσιάσεις των εκθέσεων. Επειδή δεν, έχουμε, δεν θα έχουμε εκθέσεις μέχρι το 2018, θα πρέπει να υπάρξει ένα έργο ενημέρωσης των πολιτών, των ενδιαφερόμενων χωρών, εξηγώντας τους ότι αυτό δεν θέτει να αμφιβόλο την υποψηφιότητα των χωρών αυτών. Και θα πρέπει να ε, φανταστούμε για έναν ισδά βάθος διάλογο με τις χώρες αυτές, απουσία ακριβώς των εκθέσεων αυτών, ούτω ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κατάστασης αυτής της χώρας. Γιατί η κατάσταση εξελίσσεται με καλά νέα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνα ε, υπέβαλε μια έτσι υποψηφιότητα για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ένα μη καλό νέο από την άλλη, ε, η Τουρκία εγώ διαβιώνω κατά πόσο η Τουρκία συνεχίζει να πληρεί τα κριτήρια της ε, Κοπεχάγης. Ε, γιατί η Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, θα υπάρξει μια νέα θετική έκθεση για αυτή τη χώρα. Από την άλλη έχουμε όλη επίγνωση των δυσκολιών. Είχαμε ένα παράνομο δημοψήφισμα στην Σερβία και επίσης μια παρέμβαση της Ρωσίας η οποία απροκάλυπτα υποστηρίζει αυτό το δημοψήφισμα. Ε, είχαμε τοπικές εκλογές οι οποίες ε, χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες εντάσεις. Ε, χτες καλέσαμε τον πρόεδρο συνάντηση της ΑΘΕΤ και θα ήθελα και πραγματικά χαιρετίζω την ε, προσπάθεια να υπάρξει ένας ε, πολιτικός διάλογος υψηλού επίπεδου με τις ενδιαφερόμενες ε, χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, τέσσερις σύντομες παρατηρήσεις. Κύριε Πίτροπε, καταρχήν θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για την καλή συνεργασία και εμείς από την πλευρά μας. Θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία εάν δεν έπρεπε να διαβάσουμε στην, χρειαζόταν να διαβάσουμε στη Frankfurter Allgemeine τι ε, μας περιμένει. Ε, όσον αφορά την ε, Αλβανία, έχω την, συμφωνώ με εσά. συνέβησαν πολλά τα τελευταία χρόνια. Όλοι όσοι συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο αλλά και η κυβέρνηση έκαναν αρκετές μεταρρυθμίσεις ή τουλάχιστον τις προετοίμασαν ε, νομοθετικά. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα και αν τώρα ξεκινήσει πράγματι η εφαρμογή, ε, τότε έχετε δίκιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ξεκινήσει η διαπραγματεύση το 2017. Έχετε δίκιο. Ελπίζω να συμβεί αυτό το ταχύτερο δυνατό. Δεύτερον, όσον αφορά τη Μακεδονία, μια φράση. Η Μακεδονία μπορεί να αποδείξει ότι ε, θέλει να έρθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μέσω κανονικών ε, εκλογών και ελπίζω οι πρόεδροι των κομμάτων οι οποίοι το βλέπουν έτσι να το ε, σε συμφωνία με τις, ε, σύμφωνα με τις συμφωνίες του Ιουλίου, αλλά και με ξεκάθαρη υποστήριξη ε, των, της εισαγγελία και ή δυνατόν να υπάρξει και μια διεύρυνση της εντολής τους ούτω ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Ε, τρίτο για την Τουρκία, μόνο μια φράση. Ναι, παραμένουν ε, οι εταίροι μας, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπερτέρω διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις στη βάση των κριτηρίων της Κοπενχάγης έχουν ένα νόημα και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο και η τουρκική κυβέρνηση από την δική της πλευρά ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η κατάσταση αλλάζει ραγδαία. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις, το Brexit, το μεταναστευτικό, η άνοδος των λαϊκιστικών κομμάτων, η εξάπλωση του ISIS στη Λιβύη κλπ. και οι αμερικανικές ε, εκλογές ε, τεράστιες αλλαγές με τις οποίες, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά και θα πρέπει και ενδεχομένως θα μπορούμε να εμπιστευόμαστε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μελλοντικά αν απομακρυνθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Επίσης αυτό το οποίο γίνεται στη Ρωσία και θεωρώ ότι οι ανισχύσεις της Ουκρανίας είναι εύλογες εναντί του ε, Πούτιν ή ο, η συμπεριφορά του Ερντογάν ε, στην ε, Τουρκία και αυτή μια πηγή ανησυχίας. Ε, Παρ' όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά ε, συνεχίζω να πιστεύω το ECR και το Κοινοβούλιο υποστηρίζουν τη διαδικασία της διεύρυνσης. Τώρα, όσον αφορά το Μαυροβούνιο που εγώ είμαι εισηγητής, εδώ έχουμε θετικές εξελίξεις και χαιρετίζω τις ε, εκλογές τον περασμένο μήνα. Είδα την ε, σχετική έκθεση, η οποία είναι θετική. Ε, υπάρχουν κάποια ελάσσονα θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε και απογοητεύτηκα χθε με κάποιες αντιδράσεις του Κοινοβουλίου γιατί ε, όσο ενισχύεται η, δημοκρατία εκεί θα πρέπει να αποδεχθούμε και την ενίσχυση της αντιπολίτευσης. Και θα ήθελα... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Τζουκάνοβιτς. Ε, και τέλος θα ήθελα να πω ότι το Μαυροβούνιο έχει ανοίξει τα τέσσερα κεφάλαια, δύο έχουν κλείσει προσω... προσωρινά. Thank you. I would like to start with by saying thank you, uh, Commission. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε Χάν για τη δέσμευσή σας, για την ενεργή σας συνεισφορά, για την άσκηση πίεσης την οποία κάνετε έτσι ώστε η πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι μία από τις πολιτικές μας, μία από τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Ελπίζω ότι η σύσσωμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει την επιταγή σας ε, προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να σχολιάσω και τη θέση του Συμβουλίου ε, για το μέλλον. Ελπίζω και το Συμβούλιο να σας ακολουθήσει. Πιστεύω επίσης ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι η Ευρώπη πρέπει να μεριμνήσει περισσότερο για τη δική της ευημερία σταθερότητα και ανάπτυξη. Για τη Μακεδονία, για το θέμα αυτό είμαι εγώ εισηγητής, θα ήθελα να πω ότι όλα εξαρτώνται από τις εκλογές του Δεκεμβρίου. Και ως προς τη συμφωνία και τα έγγραφα που έχουν δεχτεί, έχουν δεχτεί όλα τα μέρη τα τελευταία δύο χρόνια, πρέπει όλα αυτά να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Κύριε Χάν, στις 28 Οκτωβρίου 19 ε, οικογένειες, ελληνικές, οικογένειες ελληνικής μειονότητας έλαβαν ειδοποιητήρια κατεδάφιση των σπιτιών τους. Επειδή μας είπατε ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτή τη χώρα, πιστεύετε ότι η στάση της Αλβανίας συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντιμετώπιση των μειονοτήτων. Συνιστούν ή όχι αυτές οι ενέργειες παραβίας των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των μειονοτήτων και τι, έχετε, τι, πρωτοβουλίες θα πάρετε πάνω σε αυτό ώστε να προστατεύσετε τα δικαιώματά τους. Γιατί φύρω, Τα προηγούμενα χρόνια η χώρα βίωσε τη χειρότερη πολιτική κρίση από το 2001 παρουσιάζοντα οπισθοδρόμηση σε κέριου τομείς που αναφέρονται στα πολιτικά κριτήρια της Κοπενχάγη. Δεν πιστεύετε ότι η πολιτική ανοχή και επιβράβευση στις χώρες από την Επιτροπή μόνο ανασταλτικά λειτουργήσε μέχρι σήμερα. Και τελευταία για την Τουρκία, ε, αυτό που έχω να πω είναι ότι ελπίζω να είναι η τελευταία έκθεση που συζητάμε σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι για όσους θέλουν μια ισχυρή Ευρώπη και τις είπα ανοιχτέ στον κόσμο, όσοι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά των διακρίσεων, θα πρέπει να ε, κάνουν μια δουλειά προβληματισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Χάν. Είμαι εισηγήτρια για το Κόσοβο και συμφωνώ. Θεωρώ ότι η συμφωνία σύνδεσης και το πράσινο φως για την απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι κάτι, είναι κάτι πολύ θετικό, δύο πολύ δυνατά μηνύματα. Και παρόλο που εκτιμώ ιδιαίτερο αυτά που γίνονται, οφείλω να πω ότι τώρα το, η μπάλα είναι στο κοινοβούλιο του Κωσοβό, του Κοσφοπεδίου, για να εκπληρώσει δύο σημεία αναφοράς. Καταρχάς το προσδιορισμό του συνόρου με το Μαυροβούνιο και την απαραίτητη δράση ε, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις και τα προϋπατούμενα για το διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, μία από τις χώρες που επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αλβανία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα αυτή απέχει μακράν από το να πληρεί τις προϋποθέσεις της ε, συνθήκης Κοπενχάγης. Παρ' όλα αυτά την χάνει προστασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση της χώρας να προσπαθήσει να καλύψει αυτή τη διαφορά, κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε να καταστρέφει τις ε, σχέσεις καλής γειτονίας που οφείλει και υποχρεούται να έχει με την Ελλάδα. Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός της χώρας προέβη σε μια ανεξήγητη και απαράδεκτη επίθεση κατά της Ελλάδος, ένα πολιτικό παραλήρημα για το οποίο δεν υπάρχει, υπήρχε λόγος να γίνει. Εξέφρασε επεκτατικές βλέψεις κατά της χώρας και επιπλέον προσέβαλε και την ιστορία της χώρας. Αυτή λοιπόν είναι η πρόοδος που παρουσιάζει η Αλβανία σύμφωνα με εσά. Πρέπει να διακοπούν άμεσα οι ενταξιακές συνομιλίες μέχρι ο πρόεδρος okay. της χώρας να ορθοφρονήσει.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 Κύριε Πρόεδρε, να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Χάν για την εξαιρετική δουλειά που έκανε από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από δύο χρόνια. Νομίζω ότι στέλνετε σαφέστατα το μήνυμα ότι η διεύρυνση είναι υψηλή προτεραιότητα, ψηλά στην ημερήσια διάταξη και στον κατάλογο προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συγχαρώ για το άνοιγμα των πρώτων τεσσάρων κεφαλαίων ε, σε σχέση με την προσχώρηση τη Σερβία. Ε, για την οικονομία, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνησή του στη Σερβία πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν απασχόληση, να δημιουργήσουν ανάπτυξη, να ε, ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, υιοθετούν οικονομικέ μεταρρυθμίσει για να ενισχύσουν το φιλικό περιβάλλον, περιβάλλον φιλικό προ τι επιχειρήσει σε αυτή τη χώρα και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Η καλή περιφερειακή συνεργασία είναι απαραίτητο στοιχείο έτσι ώστε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων να πλησιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θετική προσέγγιση τη Σερβία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη μεταναστευτική κρίση και η συμφιλίωση γενικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι κάτι το ιδιαίτερο ευ ευκταίο και ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ. On Turkey. It's become, unfortunately, the top jail... Δυστυχώς ε, τίθεται το θέμα Dismissed 35.000 arrested. Ε, έχει τεθεί θέμα και για την ελευθερία του τύπου, έχουν υπάρξει χιλιάδες συλλήψεις, διώκεται η κουρδική μειονότητα. Ε, εδώ και τρία χρόνια ξεκίνησε αυτή η παλινοδία στην Τουρκία, έχει οξυνθεί τον τελευταίο καιρό. Εμείς σαν πολιτική ομάδα θέλουμε η Τουρκία να αγκυρωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Άγκυρα κλείνει την πόρτα, δεν τον κλείνουμε εμείς την πόρτα. Λοιπόν, σχετικά με τη θανατική ποινή, αν υπάρξει επαναφορά της θανατικής ποινή, προφανώς θα ασφαλιστεί η πόρτα και η δική μας, αλλά ακόμα και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει επαναφορά της δημοκρατίας στην Τουρκία. Α, αν δεν γίνει αυτό, τότε η απάντησή μας είναι αρνητική. Μια ερώτηση στον Επίτροπο. Ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες ε, της έκθεσης αυτής των 100 σχεδόν σελίδων που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, ήθελα να σας ε, ρωτήσω αν ε, έχετε λάβει υπόψη σας τις επισημάσεις που για πάρα πολύ καιρό σας έκανα ότι, και έχουν γίνει τώρα επισημάνσεις και πολλών Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι με την επίλυση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και με πολιτική και αριθμητική ισότητα, για να λειτουργήσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα πρέπει να το θέλει η Τουρκία και η οποιαδήποτε απόφαση της νέας, του νέου μορφώματο θα είναι προ το συμφέρον τη Τουρκία και θα εκφράζει τη βούλησή της αντιλαμβάνεστε ότι έστω και αν σταματήσετε τις ενταξιακέ διαδικασίες είναι ως να βάζετε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πίσω πόρτα με αυτή τη λύση που βιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ανθρώπινα δικαιώματα του Κυπριακού λαού. Αντιλαμβάνεστε πόσο άδικο είναι αυτό που επισυμβαίνει αυτή τη στιγμή και θέλετε να στηρίξετε μια λύση που δεν θα επιτρέπει στους Κύπριους στην πλειοψηφία, στη μεγίστη πλειοψηφία να εκφράζει την άποψή τη. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Ωραία. Ε, όσον αφορά τα συμπεράσματα του Επιτρόπου Χάν ε, για την ε, Τουρκία και ήδη υπόθηκε από τον κεφαλή της ομάδας μας ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεύτερον, ό,τι και να συμβεί, από την άλλη η Τουρκία είναι σημαντικός γείτονας, σημαντικός εταίρος. Δεν μου αρέσει αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί, γίνεται σε μια κλίμακα ε, την οποία ε, απευχόμαστε όλοι. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία βρίσκεται εδώ, δεν μπορούμε να την απομακρύνουμε από τη θέση της. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Υπάρχει κάποια βάση να γίνουν κάποιες συνομιλίες με τις λογικές δυνάμεις που υπάρχουν στην ε, Τουρκία. Κατά την άποψή μας η Τουρκία βρίσκεται σήμερα σε ένα τόσο βαθύ διχασμό που δεν προϊονίζεται τίποτα καλό ούτε για την ίδια ούτε δυστυχώ για τι χώρε που την περιβάλλουν ή συνεργάζονται μαζί τη. Το ερώτημα που μπαίνει είναι πώ προχωράμε, κύριε Χάν. Περιγράψετε πολύ καλά την εικόνα, όμως νομίζω ότι απουσιάζει ε, ο μοχλός που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν έχει απέναντι στην Τουρκία. Και αν υπάρχει αυτός ο μοχλός, πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει. Η αντίδραση για τη σύλληψη του κυρίου Ντεμιρτάζ είναι υποτονική. Κατά την άποψή μου δεν αρκεί να καταγγέλλεται με τον πιο σφοδρό τρόπο η σύλληψη αυτού του ανθρώπου, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι περισσότερο. Και κλείνω με το Κυπριακό ρωτώντα τον κύριο Χάν εάν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση πέραν από ευχέ τη Κομισιόν και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για επίλυση του Κυπριακού. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ως πράσινοι είμαστε πολύ υπέρ της διεύθυνσης αλλά βεβαίω υπάρχουν στιγμέ που πρέπει κανεί να σκεφτεί κατά πόσο βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Και στην περίπτωση τη Τουρκία θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του τι είναι ο Ερντογάν και τι συνιστά τη δημοκρατική Τουρκία. Και εγώ βεβαίω είμαι στο πλευρό τη δημοκρατική Τουρκία. Ενώ ο Ερντογάν ε, δεν ανήκει εκεί ε, και κάνει, οδηγεί τη χώρα σε μια σαφή οπισθοδρόμηση. Δεν κατανοώ πώ μπορούμε να συνεχίσουμε να εξαρτώμεθα από τον Ερντογάν όσον αφορά το μεταναστευτικό. Δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να επανισάγει την θανατική ποινή. Θα πρέπει εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη μας και το μερίδιό μας σε αλληλεγγύη με τους μετανάστες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εξαρτώμαστε από τον Ερντογάν και τις πολύ ασαφείς επιθυμίες του για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι θέλει η Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Είναι αυτός ο, εκείνος ο οποίος κλείνει την πόρτα, του, ε, την πόρτα σε εμά, δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς που κλείνουμε την πόρτα στην Τουρκία. E Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, αναρωτιέμαι και θέτω και το ερώτημα στους συναδέλφους. Τι άλλο πρέπει να γίνει στην Τουρκία επιτέλους έτσι ώστε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που θα έπρεπε να είχε κάνει εδώ και καιρό. Δηλαδή να δώσει ένα οριστικό τέλος στις σχέσεις μας. Ή σε, εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη ε, διαπραγματευτική διαδικασία. Ε, τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι όσοι ήταν απεσιόδοξοι είχαν δίκιο. Εμεί ανέκαθεν το λέγαμε και από την αρχή των διαπραγματεύσεων με αυτή τη χώρα. Μια χώρα η οποία και από πολιτιστική σκοπιά και από πολιτισμική σκοπιά και από γεωγραφική σκοπιά δεν αποτελεί μέρο τη Ευρώπη. Είναι μια ξένη χώρα προ τη δική μα δημοκρατική κουλτούρα. Είναι μια χώρα η οποία στρατιωτικά επίση κατέχει ένα μέρο μια ευρωπαϊκή χώρα. Μια χώρα που είναι μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η πολιτική μας είναι αδύναμη, αυτό θα είναι πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω την παρουσίαση του Επιτρόπου Χάν είναι σαφέστατα ότι ε, είναι σαφές από τα σχόλιά του ότι η διαδικασία διεύρυνσης είναι συνεχής και το ευρωπαϊκό όραμα θα ολοκληρωθεί μόνο όταν η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων προσχωρήσει πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι η διαδικασία διεύρυνσης ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε μια πιο σταθερή και ευημερούσα Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν και άλλες χώρες να κάνουν τη δική τους δουλειά, το, να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, να έχουν δημοκρατική λειτουργία και να ενθαρρύνουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Έχω όμως δύο παρατηρήσεις να κάνω. Συζητούμε τη διεύρυνση και το πακέτο διεύρυνσης και την έκθεση αναχώρα. Δεν είναι καλή ευκαιρία ε, για να σπρώχνουν οι διάφορες χώρες ξεχωριστά τα δικά τους συμφέροντα έναντι της μίας ή της άλλης υποψήφιας χώρας. θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και να επιδείξουμε πνεύμα ευγενούς αγαστή συνεργασίας με τον Επίτροπο Χάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Εμείς χρειαζόμαστε τα Δυτικά Βαλκάνια περισσότερο από ποτέ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και εμείς και αυτοί. Τα πράγματα όμως δεν πηγαίνουν ε, κανονικά όπως θα έπρεπε. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ό,τι είπατε. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης ή πληρώνονται πάρα πολύ λίγα. Οι νέοι εγκαταλείπουν τις ε, χώρες τους, αυξάνεται ο εθνικισμός. Θέλω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρώσει την προσοχή της ιδιαίτερα στις μελλοντικέ εξελίξεις και την ανάπτυξη της Βοσνίας Ευζεγοβίνης. Θα ήθελα επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη από πλευρά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών του Κωσυφοπεδίου. Και τέλος, θα πρέπει να αλλάξουμε ε, την, την, τις ανακοινώσεις μας, τη δημοσιότητα των προσπαθειών που κάνουμε. Να μην λέμε μόνο ανοίγουμε ή κλείνουμε κεφάλαια, να πούμε περισσότερα και να εξηγήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πολύ καλές προσπάθειες που κάνετε για τα Βαλκάνια, για το θέμα της ατζέντα για τη συνδεσιμότητα, για τους διαδρόμους τους μεταφορικούς. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν αρκετές ομοιότητες, πρέπει να προχωρήσουν στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και είναι και αλληλοεξαρτημένες μεταξύ τους. Γι' αυτό τα κοινά προγράμματα για τις χώρες αυτές παίζουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η ερώτησή μου λοιπόν και πρόταση προς τον Επίτροπο είναι η εξής. Ε, θα υπάρξουν ε, περαιτέρω νέα κοινά προγράμματα στον τομέα έστω και της δικαστικής εξουσίας ή της δημόσιας διοίκησης, κοινά προγράμματα για όλες τις χώρες. Uh, Συγγνώμη κύριε. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω τον Πέτρο Χάν για την συνεργασία σας και τις προσπάθειες που κάνετε τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Όπως όλοι διαπιστώσαμε σήμερα το πρωί, ο κόσμος μεταβάλλεται ραγδαία. Ε, νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε οι περισσότερες χώρες να πρέπει να παράσχουν συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Οι εκθέσει για τα Δυτικά Βαλκάνια ε, ε, διαπιστώνουν κάποιες εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αδυναμίες στην διοίκηση και ψηλά ποσοστά ανεργίας. Από την άλλη η περιφερειακή συνεργασία έχει βελτιώσει ε, είμαι ευτυχής ε, που θα συνεχιστεί η διεύρυνση χωρίς την εσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων η Ευρώπη δεν θα, είναι ενωμένη και αναμένω με ανεπομονησία την ε, γνωμοδότηση του Επιτρόπου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και ελπίζω ότι θα είναι βιώσιμη η ανάπτυξή Δεν θα αναφερθώ στο ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε μια πέραντη φυλακή όπου φυλακίζεται όχι όποιος εκφράζει τη διαφωνία του, αλλά όποιος σκέφτεται διαφορετικά από τον κύριο Ερτογάν. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε να διεξάγονται συνομιλίες στην Ελβετία για επίλυση του Κυπριακού μεταξύ του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ηγέτη των Τουρκογυπρίων και η Τουρκία είναι παρούσα κατά έμμεσον τρόπο. Δεν πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο ούτως ώστε η λύση να είναι συμβατή με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην δίνει στην Τουρκία το δικαίωμα να έχει λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο Χάν για το έργο του. Μια σύντομη παρατήρηση για τη Σερβία. Χαίρομαι διότι η έκθεση για τη Σερβία περιλαμβάνει πολλές θετικές παρατηρήσεις για διάφορα πεδία. Ως προς τα δικαιώματα των ε, ε, εθνοτικών μειονότητων, αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά ενδιαφέρον για όλους εμάς και θέλω να σας ενημερώσω ότι η Διακοινοβουλευτική Ομάδα για τις Εθνοτικές Μειονότητες στην τελευταία συνεδρίαση στο Στρασβουργό είχε τη χαρά να ακούσει τον αρμόδιο Σέρβο Υπουργό που παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τις εθνικές μειονότητες της χώρας και τι δράσει που αναλαμβάνει η σερβική κυβέρνηση για την εφαρμογή του σχεδίου δράση. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση το έχει θέσει αυτό ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων τη. Δεν έχουμε την ακριβή διατύπωση της έκθεσης ακόμα, δεν έχει δημοσιευθεί επισήμως. Θα ήθελα όμως ε, λίγα σχόλια από δική σας πλευρά, κύριε Επιτρόπη, πώς αξιολογείτε αυτό το σχέδιο δράσης και την εφαρμογή του. Ευχαριστώ. Ο εθνικισμός, ο λαϊκισμός στην Ευρώπη, αντίστοιχα φαινόμενα στη ΣΥΠΑ, στον κόσμο, μας οδηγούν να καταδικάσουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που καταστρέφουν θέσεις απασχόλησης, απορριθμίζουν τον κόσμο και τροφοδοτούν ε, βεβαίως τον Τραμπ, τον Ερντογάν, πολιτικούς τέτοιου τύπου όπως και τον επικεφαλής της ΚΑΓΕΜΠΕ Πούτιν. Πρέπει να επανέλθουμε στις ευρωπαϊκές αξίες και αυτό δεν ισχύει με την Τουρκία υπό τον Ερντογάν σήμερα. Ο Ερντογάν είναι αυτό που κλείνει την πόρτα, είναι αυτό που καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και εγκαταλείπει την εφαρμογή του κράτου δικαίου. Πρέπει να παγώσουμε τι διαπραγματεύσει και πρέπει να εμπλακούμε ακόμα περισσότερο ενεργητικά σε συνεργασία με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία για να απευθύνουμε έκκληση για την επαναφορά τη δημοκρατία στη χώρα αυτή. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάν για σημαντική παρουσίαση και πραγματικά για το έργο σας στα Δυτικά Βαλκάνια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια είναι προς όφελος των πολιτών αυτής της, αυτών των χωρών και προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλές, πολλές θετικές παρατηρήσεις στις εκθέσεις αυτές ε, για διάφορες χώρες ε, ε, Βεβαίω υπάρχουν περιθώρια βελτίωση σε άλλου τομεί και φοβούμαι ότι δεν συζητήσαμε αρκετά το θέμα της οικονομικής κατάστασης της περιοχής αυτής. Ε, είμαι σίγουρος ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι αναπόσπαστο τμήμα ε, του έργου μας και συμφωνώ με όσους είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδράμει περισσότερο αυτές τις χώρες, γιατί χωρίς θέσεις απασχόλησης, χωρίς εκπαίδευση των νέων στις χώρες αυτές, δεν θα υπάρξει μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, οποιαδήποτε χώρα με μη ανεξάρτητο δικαστικό σήμα ε, θα, θα πρέπει να θεωρηθεί δικτατορία στην Τουρκία βάσει των στοιχείων τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου. Η, η χώρα κυβερνάται με προεδρικά διατάγματα, δεκάδες χιλιάδες ε, αγνοούνται, φυλακίζονται ε, βουλευτές, ε, δήμαρχοι και Κούρδοι, απλώς και μόνο επειδή είναι Κούρδοι αλλά δεν περιγράφεται αυτά ως τυραννία ούτε ως δικτατορία. Το δεύτερο σχόλιο μου αφορά την Κύπρο. Η πολιτική ε, αμοιβή ε, ε, της Τουρκίας έχει αποτύχει. Τι θα γίνει με την Κύπρο. Θέλουμε η Τουρκία να παράσχει τις εγγύης. Ποιος θα προστατεύσει εμάς από τον Ερντογάν. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κατ' ουσία θα πρέπει να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αυτή η εκδήλωση εδώ, αυτή η συνεδρίαση εδώ είναι μια φάρσα. Ε, μαθαίνουμε από τον τύπο προηγουμένως ε, τι ε, περιέχει η έκθεση της Επιτροπής. Και αυτό το οποίο διαβάζω στον τύπο για την Τουρκία αυτό αντανακλά την άνοδο στην εξουσία ενός δικτάτορα. Δεν ε, τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου δεν υφίσταται πλέον, ούτε η δημοκρατικότητα, ούτε η δημοκρατία. Πού είναι εδώ η, επιτροπή της, η πρώτη επιτροπή, πού είναι η πολιτική αξιολόγηση, πάβει η Κομισιόν να λειτουργεί ως θεματοφύλακα των συνθηκών. Βεβαίω ε, Συμφωνώ, ναι, θα πρέπει να ε, παραμείνουμε σε διάλογο με την Τουρκία, γιατί αυτό το οφείλουμε στους αθώους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν θα έπρεπε να εκφράσει πιο ρητά τη δική της τοποθέτηση. ευχαριστώ πολύ κύριε Χάν για τη δουλειά, για τη δουλειά σας. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Είμαι αρμόδιο εισηγητή για το θέμα και χαίρομαι για τι θετικέ εξελίξει, διότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε τέλμα η κατάσταση ε, στη χώρα αυτή και τώρα ο κόσμο έχει ελπίδε για ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον. Πολλά μένει να γίνουν, οι εντάσει έχουν επιδεινωθεί μεταξύ, τους, ε, μεταξύ των Σερβοβόσνιων και των Κροατοβόσνιων και ε, το δημοψήφισμα των φιλεγόμενων στη Ρεπούμπλικα Σερβσκά. Επίσης γνωρίζουμε ότι η σταθερότητα, η αστάθεια στα Βαλκάνια ήταν ε, επικίνδυνη για τη διεθνή σταθερότητα και η ειρήνη. Πρέπει να είμαστε αληθινοί και όχι ουδέτεροι. Διάφορες δράσεις παραμένουν χωρίς κυρώσεις. Και αν ε, μείνουμε απρακτοί θα έχουμε νομική αναρχία και περαιτέρω αποδόμηση. and this way practically everyone who was on this list had the chance to speak. And thank you very much for all. Όλοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, νομίζω, που είχα στον κατάλογο των ομιλητών. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για τις ε, παρεμβάσεις σας. Θα ήθελα επίσης να, ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω που τηρήσατε τα χρονικά περιθώρια. Και, γιατί και εγώ συνηθίζω να τηρώ τους κανόνες του παιχνίδιου και οι κανόνες αυτοί ε, προβλέπουν καταρχήν ότι εγώ κάνω μια παρουσίαση εδώ και στη συνέχεια δίδω μια συνέντευξη τύπου. Ε, αλλά ε, θα υπάρξουν και στο μέλλον αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε την κατάσταση στις διάφορες χώρες. Το γεγονός ότι η επόμενη έκθεση θα, εκπονηθεί, θα είναι έτοιμη το 2018 καθορίζει το χρονοδιάγραμμα ε, το οποίο θα πρέπει να μετατεθεί για, από το φθινόπωρο για την Άνοιξη. Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, θα ήθελα να δείξετε κατανόηση ότι δεν μπορώ να επιστέλθω σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές άλλε δυνατότητες. Γι' αυτό θα περιοριστώ σε ορισμένε παρατηρήσεις γενικής φύσεως. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κυρίως για την επισήμανση ότι στα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για την οικονομική ε, ανάπτυξη. Είναι η περιοχή με, τη, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεργία των νέων. Ε, έχουμε πολύ μεγάλη διαρροή εγκεφάλων εδώ και δυστυχώς είναι τα πιο δυναμικά στοιχεία μιας κοινωνίας αυτά τα οποία φεύγουν και οι νέοι άνθρωποι ε, στα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να έρθουν στο επίκεντρο της προσοχής μας και της ενισχυμένη συνεργασίας ε, στο επίπεδο των ανταλλαγών, όχι μόνο των ακαδημαϊκών ανταλλαγών, αλλά και μεταξύ ανθρώπων που κάνουν κάποια μαθητεία, ε, ούτως ώστε να υπάρξει δυνατότητα να συγκεντρωθούν εμπειρίες και να υπάρξει και μια ανταλλαγή εμπειριών, ούτως ώστε οι νέοι ε, και που απασχολούνται στην ε, δημόσια δίκηση για παράδειγμα να κάνουν κάποιες εμπειρίες στη Γαλλία επί παραδείγματι και να μπορέσουν επιστρέφοντας στις χώρες τους να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις. Ε, βεβαίως η οικονομική εξέλιξη είναι σημαντική ε, και βεβαίως θα θέσει τις ε, προϋποθέσεις για μια εξέλιξη του κράτους, κράτους δικαίου γιατί θα βρείτε ε, διεθνείς επενδυτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόνον εφόσον στις χώρες αυτές υπάρχει μια καλώς λειτουργούσα δικαιοσύνη και μια σωστή νομοθεσία. Αλλιώς δεν είναι κανείς ε, διατεθειμένος να ρισκάρει τα χρήματά του εφόσον είναι σαθρά τα ε, συστήματα της ε, δικαιοσύνης. Θα ήθελα ωστόσο να σας παρακαλέσω και να δείξετε μια κατανόηση όσον αφορά την εξέλιξη στις διάφορες χώρες εμείς ε, είμαστε ε, υπεύθυνοι για, την, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εδώ θα έβαζα θετικό πρόσημο ε, βεβαίως αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ε, εδώ και εκεί κάποια ελλείμματα τα οποία δεν θα πρέπει να αρνηθούμε όσον αφορά για παράδειγμα την, ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων που αποτελούν στοιχείο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε με τις αντίστοιχες κοινωνίες και ελπίζουμε να εξελιχθούν προς τη σωστή κατεύθυνση οι κοινωνίες των χωρών αυτών γιατί το ζητούμενο δεν είναι να ευρεθούν αυτά μόνο στους νόμους, να διατυπωθούν μέσω νόμων, αλλά θα πρέπει οι νόμοι αυτοί να εφαρμοστούν. Γιατί ακριβώς ε, πρόκειται για μια διαδικασία και αυτό θα πρέπει να το θέσουμε στο επίκεντρο των ε, προβληματισμών μας. Δεν πρόκειται για μια υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου εκ μέρους των χωρών αυτών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια εξέλιξη των χωρών αυτών ε, στις, ε, στην κατεύθυνση αυτή. Ε, ο τρόπος που εμείς δίνουμε τα χρήματά μας και ποια προγράμματα εφαρμόζονται και εδώ ε, θα πρέπει να υπάρξει μια πιο έντονη ορατότητα των ε, επενδύσεών μας ε, σε σχέση με τον απλό πολίτη. Γιατί κάνουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την υποστήριξη του προπολογισμού κλπ. Είμαστε με απόσταση ο μεγαλύτερος δωρητής στην περιοχή αυτό, αλλά ως γνωστόν αυτό δεν προσλαμβάνεται παρκώς από τους πολίτες των χωρών και βεβαίως εδώ θα πρέπει να κάνουμε ε, κάποιες ε, βελτιώσεις ε, στην ορατότητα των στόχων μας, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε ταυτόχρονα και την επικοινωνία με τις χώρες αυτές, επιδεικνύοντας μεγαλύτερο ζήλο σε αυτή την, ε, και δέσμευση στην επικοινωνία αυτή με τις χώρες αυτές. Αλλά βεβαίω πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ε, ένα φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό, γιατί πολύ συχνά οι τοπικές ε, κοινωνίες δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βάζουν στην άκρη γιατί τρέπονται. Ε, και αυτό το ξέρω και από χώρες εντός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που συχνά ε, καταφεύγουν σε αυτή την πρακτική. Το ξέρω από τη δική μου εμπειρία στο παρελθόν. Οι χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει λοιπόν να και θα πρέπει να, αναλάξουμε την κατάσταση αυτό, αυτή. Όσον αφορά την Τουρκία, νομίζω ότι ε, είμαστε αρκετά ξεκάθαροι στην έκθεσή μας, αλλά αναμένω στη βάση αυτής της έκθεσης όχι μόνο από τη δική σας πλευρά και υπήρξατε πολύ σαφείς, αλλά και στο επίπεδο των χωρών μελών αναμένω να λάβει η χώρα μια επί της ουσίας, συζήτηση την επόμενη Δευτέρα στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών θα υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα και ελπίζω να υπάρξει μια ακριβής καταγραφή της κατάστασης ούτως ώστε και εμείς ε, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εις βάθος συζητήσεις με τους Τούρκους εταίρους μας. Γιατί είναι αδιαφυσβήτητο και το είπατε άλλωστε και εσείς ότι η Τουρκία υπό την παρούσα τουλάχιστον κυβέρνηση ε, αποκλίνει όλο και περισσότερο από την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας να μην χάνουμε από το μυαλό μας ότι υπάρχουν 80 εκατομμύρια Τούρκοι ε, πολίτες οι οποίοι και αυτοί θέλουν να έχουν μια προοπτική και εδώ θα πρέπει να αναλάβουμε ένα μερίδιο ευθύνη, δικής μας ευθύνη, καθώς και ένα μερίδιο ευθύνη για όλους εκείνους οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές και οι οποίοι, τον οι θέλουν να το δικαίωμα στη διεξαγωγή μιας δίκης δίκης. Και θα ήθελα να εξαντλήσω τις δυνατότητες των διμερών επαφών ε, να μπορέσουμε να κάνουμε μια παρατήρηση της διεξαγωγής αυτών των ε, διαδικασιών ούτω ώστε να γίνουν σύμφωνα με τι αρχέ του κράτου δικαίου. Αλλά θα πρέπει να πω ότι η Τουρκία μέχρι στιγμή δεν απάντησε στη δική μα πρόταση να υπάρξει παρακολούθηση και υποστήριξη από τη δική μα πλευρά ε, του τρόπου με τον οποίο θα διεξαχθούν όλε αυτέ οι δίκε. Και ε, ενώ θα ήταν ισόφελος τη χώρα να τεκμηριώσουμε ότι πράγματι ε, συνάδουν οι διαδικασίες αυτές με τις αρχές του κράτους ε, δικαίου. Όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα, και εδώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε ότι πρωτίστως πρόκειται για τους ίδιους τους ανθρώπους, για την τύχη αυτών των ανθρώπων, ε, τους μετανάστες, για τους οποίους θέλουμε να εξασφαλίσουμε τις συνθήκε συνθήκες διαβίωσης στα στρατόπεδα αλλά και στο δημόσιο χώρο όχι μόνο η στέγαση και η διατροφή, αλλά και η εκπαίδευση ε, να εξασφαλίζεται, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί το ταχύτερο δυνατό να επιστρέψουν στις αιστείες τους στη Συρία. Και αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι για δικό μας, δικό μας όφελος και θα έπρεπε ε, ε, να δούμε ότι η συνεργασία με την Τουρκία είναι για το δικό μας συμφέρον. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να κλειστούμε από την Τουρκία. Υπάρχει μια συμφωνία από τη μία και την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η μορφή της συνεργασίας και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τομείς όπου τα πράγματα δεν λειτουργούν και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς τους τομείς και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τη δική σας ε, ομάδα όπως και την ε, δική μας είμαστε πολιτικά ηθήνοντες αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε το επιτελείο μας και θα έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τόσο το δικό σας και το δικό μας επιτελείο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. Αυτή είναι η αρχή μιας διαδικασίας που θα πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο.